la proposition du président, euh, Μετά από πρόταση του Πρόεδρου Λάμπερτς και τις κατηγορίες του που ήταν δίκαιες, ότι καθυστερώ, κήρυσε την έναρξη των εργασιών μας. Ο ένας εισηγητής μας έφτασε, ο άλλος δεν θα έρθει σήμερα. Λοιπόν, έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται. Έχετε επίση καταλάβει ότι έχουμε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα, πιο σημαντική από ό,τι συνήθω, που αποτελείται από δύο εντελώ διαφορετικά μέρη. Πρώτον, θα έχουμε την παρουσίαση από τον κ. Κοφόντ του σχεδίου έκθεσης που Ακπώνησε μαζί με τον κύριο Τόιρ και θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τους σκιώδεις εισηγητές από όλε τις πολιτικές ομάδες, αλλά και άλλους που θα πάρουν το λόγο εδώ. Ο εισηγητής εννοείται ότι θα πάρει το λόγο και στο τέλος για να κλείσει αυτή η συζήτηση, καταλήγοντας σε συμπεράσματα και σε πολιτικά μαθήματα, τα οποία εξάγονται από τη συζήτησή μας. για τροπολογίες που ενδεχομένως μπορούν να υποβληθούν ακόμα στην έκθεση. Στο δεύτερο μέρος συνεδριάζουμε μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Με τους συντονιστές αποφασίσαμε να έχουμε από κοινού ακρόαση, εκείνη και εμείς, όσον αφορά τις ε, συνέπειες για τις υπονάπτυξη χώρες των ε, φορολογικών σχεδιασμών και της φοροαποφυγής. Συνέπειες επιθετικών φορολογικών πρακτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτός είναι ο τίτλος. Λοιπόν, ανακοινώσεις του Πρόεδρου έχουν γίνει γραπτά. Να κερδίζουμε χρόνο, δεν θα τις επαναλάβω. Θέλω όμως να επενθυμίσω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της έκθεσης αυτής. Ότι έχετε στη διάθεσή σας ή έχουμε στη διάθεσή μας από την 11η Μαΐου στα αγγλικά το σχέδιο έκθεσης. Από χτες μάλιστα έχουμε και όλες τις γλώσσες. 24 του μηνός έχουμε την ανταλλαγή απόψε και την παρουσίαση της έκθεσης. Και όσον αφορά την προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, είχαμε προβλέψει την 27η Μαΐου. Πιστεύω όμως ότι δεν φτάνει. Είναι πολύ σύντομα. Και γι' αυτό προτείνω να υπάρξει μια μικρή αναβολή για την 3η 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Τότε είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ξέρω ότι τη χρειάζεστε αυτή την παράταση. Και εγώ θα ήθελα να έχω το χρόνο να διαβάσω όλες τις λεπτομέρειες στο κείμενο και να λάβω υπόψη μου και τόσα θα υποθούν εδώ. Από τις 11 Μαΐου και μετά υπήρξαν και άλλες εργασίες. Λάβαμε γνώση νέων εγγράφων. Σήμερα το πρωί γίνεται μια σημαντική συνάντηση συντονιστών και σκιωδών επί των εγγράφων αυτών. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή. Στείλαμε επίσης αντιπροσωπεία τις οποίες εγώ ηγήθηκα μάλιστα, στην Ουάσιγκτον. Πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή αυτή. Και από αυτού θα συζητήσουμε. Είχαμε εκεί επαφές και με τις Αμερικανικές αρχές υπεύθυνε για αυτά τα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών. Είχαμε επαφές επίσης με το Κογκρέσο, αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα και με τα δύο πολιτικά κόμματα και φυσικά συναντηθήκαμε και με πανεπιστημιακούς, με την Παγκόσμια Τράπεζα, την Oxfam και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όλα αυτά θα οδηγήσουν βέβαια σε τροπολογίες, σε επιπλέον τροπολογίες, γι' αυτό και χρειαζόμαστε την παράταση. Προτείνω λοιπόν, α, ο Πίτερ Σίμον θέλει ένα σχόλιο πριν δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, σωστά. Πίτερ, έχεις το λόγο. Ζήτησα τον λόγο γιατί ήμουν στην συζήτηση των συντονιστών για το θέμα των εγγράφων και την πρόσβαση στα έγγραφα και μία παράκληση από όλους τους συντονιστές ήταν σαφής. Ακούστηκε και θα το πούν και οι συνάδελφοι της ΓΚΟΕ πως κάποια έγγραφα δεν βρίσκονται ούτε στην αίθουσα ούτε είναι από αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που η Κομισιόν τα έχει, αλλά σύμφωνα με δηλώσεις ε, της ε, ΓΚΟΕ κοστίζει πολύ να μας τα μοιράσουν. Παρακαλώ να το ξαναδείτε και παρακαλέστε να μας ε, να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Για να, έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα υπάρχοντα έγγραφα. Το δεύτερο θέμα. Μάθαμε πως είναι περιορισμένη η πρόσβαση στα έγγραφα μέχρι 15 Ιουνίου. Θεωρώ πως αυτή η προθεσμία είναι από προηγούμενη θητεία. Νομίζω καλό είναι να ε, έχουμε πρόσβαση μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Καλώς. Σημειώνω λοιπόν και θα φροντίσω τα αναγκαία ώστε να ζητήσω και πάλι επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτά και τα λοιπά τη νέα αυτή κατηγορία εγγράφων που λείπουν. Σας ευχαριστώ. Γέπε, για την παρουσίαση της έκθεσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και σε όλους τους συναδέρφους που είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και εκείνους που έχουν ήδη στείλει τις προτάσεις τους γραπτά. Όπως ε, ξέρετε, ο Μάκλ Τόιερ, ο συνεισηγητής, δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Αλλά ξέρω ότι κάποιοι από την άλλη έχουν ένα δικό του σημείωμα. Ο Τόιερ και εγώ λοιπόν, πριν πω στην ουσία και το περιεχόμενο, ο Τόιερ και εγώ ακολουθήσαμε την ίδια ανοιχτή διαδικασία με συνομιλίες, διαβουλεύσεις. Ο χρόνος βέβαια πιέζει. Το γνωρίζουμε αυτό και έχει υποθεί ξανά και ξανά. Τώρα, είναι σημαντικό με το χρονοδιάγραμμα αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας να δείξουμε όλη ευελιξία και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμβιβαστικές λύσεις. Μετά την παρουσίασή μου, επίσης προσβλέπω στις δικές σας προτάσεις και σχόλια, τα οποία θα σημειώσω πολύ προσεκτικά όλες τις τοποθετήσεις των πολιτικών ομάδων, έτσι ώστε από την Επιτροπή μας να βγει μια ισχυρή έκθεση. Να αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τους πολίτες μας, ότι ο επιθετικός ε, φορολογικός σχεδιασμός, η φοροαποφυγή είναι πράγματα παράδεκτα και είναι πράγματα που δεν θέλουμε. Η Επιτροπή μας, η ΤΑΞ και η ΤΑΞ 2 βλέπει κάποια πρόοδο, αλλά θέλουμε περισσότερη πρόοδο. Στην έκθεση αυτή λοιπόν υπογραμμίζουμε τα όσα βγήκαν από την Επιτροπή Ταξένα. Όλες, ε, όλα τα συμπεράσματα, οι αποφάσεις και τα λοιπά λαμβάνονται υπόψη, ισχύουν και με την έκθεσή μας αυτή της τάξη 2 ενισχύουμε ουσιαστικά τα συμπεράσματα της ΤΑΞΕΝΑ. Μην ξεγελιέται κανείς ότι επειδή εδώ δεν επαναλαμβάνουμε κάποιο συμπέρασμα, δεν το θεωρούμε σημαντικό, απλώς δεν θέλουμε να υπάρχει επικάλυψη και στα πάντα. Βασιζόμαστε όμως στα συμπεράσματα της πρώτης Επιτροπής. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα τμήμα που αναφέρει όλα τα στοιχεία και όλες τις έρευνες που έγιναν όσα ακούσαμε εδώ στην Επιτροπή μας και τι εξελίξεις υπάρχουν από τότε που εγκρίθηκε η έκθεση της TAX 1 και μετά. Στη συνέχεια κοιτάμε το ρόλο των φορολογικών δικαιοδοσών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό Κοιτάμε τις πατέντες που ισχύουν, τη γνώση, τα λεγόμενα boxes. Κοιτάμε επίσης τα έγγραφα της ομάδος κώδικα θεοντολογίας, το G20, g κλπ. και τις συνέπειες επίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, για τις οποίες έχουμε ακρόαση μετά. Στη συνέχεια κοιτάμε πώς θέλουμε να προχωρήσει η τάξη 2. Τώρα, δεύτερον, συνοψίζουμε τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις δράσεις της μετά από την έκθεση TAX 1. Αυτή ήταν και η εντολή εξάλλου που πήραμε ως TAX 2. Έπειτα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και αξιολογήσεις. Έχουμε έξι ανεξάρτητα θέματα για τα οποία γίνονται διάφορες συστάσεις. Φυσικά αυτό είναι και το πιο σημαντικό τμήμα της έκθεσης. Κάναμε προσπάθεια να συμπεριλάβουμε και τα όσα γραπτά μας πρότειναν οι σκιώδεις εισηγητές. Και θέλω να υπογραμμίσω πόσο μεγάλη σημασία έχουν όλα αυτά και θα αναφερθώ σε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, κυρώσεις και ένας κατάλογος, μια μαύρη λίστα για όσες δικαιοδοσίες δεν συμμορφώνονται. Πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προ αυτή την κατεύθυνση, να υπάρχει δηλαδή φορολογική δικαιοσύνη. Είναι προτεραιότητα στην έκθεσή μα να αντιμετωπιστούν οι φορολογικοί παράδεισοι. Πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, μια μαύρη λίστα προκειμένου αυτή να εγκριθεί πριν από τα τέλη του 2016. Και θέλουμε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για κυρώσει κατά των δικαιοδοσών εκείνων που δεν συμμορφώνονται ή όσο βρίσκονται στον κατάλογο αυτό στη μαύρη λίστα με κυρώσεις που μπορεί να φτάνουν ε, στο σημείο διακοπής συμφωνιών χρηματοδότησης κλπ. Είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για συμβούλους, είτε πρόκειται για τράπεζες. Συστήνουμε επίσης την ε, εισαγωγή ενός συστήματος που να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει διπλή φορολόγηση. Τη θέλουμε συνοχή φορολογική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική ε, φορολογική πολιτική που να καλύπτει τα κενά τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα και από τα οποία επεφελούνται πολύ. Στη συνέχεια, δεύτερο τμήμα είναι πατέντες, γνώση και τα λεγόμενα boxes θα επεκταθώ περισσότερο αργότερα. Χρειαζόμαστε δεσμευτικά μέτρα για να μην εποφελούνται πολλοί από αυτές τις αδυναμίες και να συμμορφωνόμαστε στις οδηγίες ώστε να μην υπάρχουν εξαιρέσεις για τις τράπεζες, για τους συμβούλους, για τους ενδιάμεσους. Είχαμε διάφορες ακροάσεις με τις τράπεζες εδώ και από τα έγγραφα του Παναμά φάνηκε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο κώδικας δεντολογίας για όλες τις συμβουλευτικέ υπηρεσίες είναι επίσης κάτι που προτείνουμε. Και μία αναλογική υποχρέωση για όλους όσοι διευκολύνουν τη μεταφορά χρημάτων σε φορολογικούς παραδείσους. Έπειτα υπάρχει το θέμα των whistleblowers, των καταλαγιόντων. Φάνηκε και από τα έγγραφα του Παναμά ότι η πίεση πρέπει να παραμείνει και στην Επιτροπή και στις χώρες μέλη, εννοείται, πάνω απ' όλα χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο για να διασφαλίσετε αποτελεσματική προστασία των καταγγελόντων. Οι χώρε μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν την νομοθεσία του έτσι ώστε να μην διώκονται δημοσιογράφοι και καταγγέλλοντε. Έτσι, στέλνουμε ένα μήνυμα και στο Λουξεμβούργο, αναφέροντας και πάλι τα LuxLeaks. Η προστασία βέβαια του απορρίτου των επιχειρήσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, να χρησιμοποιείται σαν άλοφη για να διώκονται ε, καταγγέλλοντες οι οποίοι αποκαλύπτουν αθέμητες πρακτικές. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε για να το υπογραμμίσουμε. Η ομάδα τώρα κώδικα θεντολογίας και θεσμικά ζητήματα. Υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες που αναφέρονται. Το βασικό είναι ότι υπάρχει αποτυχία αναθεώρηση τη ομάδα κώδικα διοντολογία. Οι χώρες πρέπει να προχωρήσουν. Είναι κάτι που το ζητάμε. Όπως επίσης και περισσότερη διαφάνεια. Είναι κάτι που θα επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Όσον αφορά τώρα το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται ώστε οι χώρες μέλη να μπορούν να μετρήσουν το θέμα της φορολογικής αποτελεσματικότητας και να δούνε και το θέμα της διασυνοριακής φοροαποφυγής. Έχουμε και ένα κομμάτι για την εξωτερική διάσταση. Ζητάμε από τον ΩΣΑ να ξεκινήσει με τις βέλτιστες πρακτικές και να αναφερθεί και στο BEPS 2 ε για ελάχιστες προδιαγραφές και συγκεκριμένους ε, στόχους που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα σημεία του ΠΕΠΣ. Να υπάρχει υποπτική ομάδα η οποία θα ελέγχει το έργο των ΠΕΠΣ και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει σε όλες τις εταιρικέ και εμπορικέ συμφωνίες ρήτρε χρηστής διακυβέρνησης. Καλή εφαρμογή των μέτρων ΠΕΠΣ και σεβασμό των προδιαγραφών. Εδώ, επειδή μιλάμε για την εξωτερική διάσταση, θέλουμε να βάλουμε και τις βάσεις για μια διεθνή πρωτοβουλία. Ζητάμε δηλαδή κάτι που μπορεί βραχυπρόθεσμα να μην είναι εφικτό, αλλά είναι σημαντικό, να υπάρχει ένα μητρό στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων ε, κτλ. που περνάνε από τις φορολογικές αρχές. Είναι συγκεκριμένες προτάσεις, έχουμε συζητήσει την ουσία. Αυτό όμως που θέλω να επαναλάβω είναι ότι εμείς οι δύο εισηγητές είμαστε στη διάθεσή σας. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας θα βρεθούμε ξανά και ξανά με τους σκιώδεις, με την Επιτροπή ολόκληρη για να συζητήσουμε και να ξανασυζητήσουμε την έκθεση αυτή. Έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί, να καταλήξουμε σε μια ισχυρή έκθεση. Γιατί αυτό το θέμα για μένα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να οδηγηθούμε σε δράσεις μετά από αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Σιγητά και συγχαρητήρια για το αξιόλογο έργο το οποίο ολοκληρώσατε σε συνεργασία με τον κύριο Τόιλερ. Καταλήξατε σε αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι άριστη βάση εργασία και διαμαντεύσεων, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ το τελικό κοινό εκθεσμό. Κύριο, ε, τώρα δεν είναι εκεί, αλλά η κυρία Σιλίγκουλαρ θα μιλήσει εκ μέρου του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ακριβώ θα διαβιβάσω όλα τα καλά σα λόγια. Και εξ του κύριου Τόιλερ, αν να σα τα πω στα αγγλικά. Για... Μιλήσω αγγλικά. Ε, δεν μπόρεσε να ήθελα, αλλά ήθελα να ευχαριστήσει τον ε, συνεισηγητή και τους συναδέλφους και ήθελα να σας υπενθυμίσει τα αποτελέσματα της πρώτης ειδική Επιτροπής το γεγονό πως ο συνδυασμός 28 περίπλοκων ε, φορολογικών συστημάτων οδηγεί σε παραθυράκια τα οποία εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές για φοροαποφυγή και έτσι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός όπως θα θυμάστε η τάξη 1 ζήτησε ένα δεσμευτικό ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο και μια κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Και ως πρώην σκιώδης εισηγήτρια επί του θέματος ε, και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Υπήρχαν όμως ε, διάφορα ζητήματα τα οποία δεν τα είχαμε ολοκληρώσει στην πρώτη εντολή, π.χ. η εξωτερική διάσταση αλλά και ο ρόλος των τραπεζών, ενδιαμέσων και κρατών που δεν συνεργάζονται. Αυτά είναι λοιπόν ε, τα ζητήματα τα οποία ήθελε να θέσουμε ο Μιχαήλ στην τάξη 2 και λέει τα εξής να ζητήσουμε ένα φορολογικό καθιστό στη συνθήκη να εφαρμόζονται οι φόροι ώστε να μην ε, επιβάλλεται διπλή φορολογία και επίσης να δούμε τα καθεστώτα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα patent boxes και όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς και την πρόσβαση στα έγγραφα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε πλέον πρόσβαση. Είναι περίεργο όμως το ότι αρκετά έγγραφα κάπου χάθηκαν και δεν, μπορού, δεν μπόρεσε να μας τα δώσει η Κομισιόν. Συμπερασματικά λοιπόν το σχέδιο έκθεσης βασίζεται στην έκθεση της ε, πρώτης ε, θητείας ε, της Επιτροπής μας αλλά υπό το φως των αποκαλύψεων του Παταμαναμά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει έναν τρόπο να πάει πέρα και από την εντολή της Ειδικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος προς την κυρία Γκουλάρ. Και τώρα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Όπως πάντα, μέχρι πέντε λεπτά μπορείτε να αγοράσετε πρώτη. Η τα Χίμνερ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Αλέν, θα ήθελα να αρχίσω αναφέροντας ότι βέβαια έχουμε πολλές προκλήσεις και βέβαια πρόκειται για δύσκολη έκθεση. Και επιπλέον δυσκολία νομίζω ότι προέρχεται από το γεγονός ότι μάλλον είναι πρόημο να αξιολογήσουμε τις συστάσεις της πρώτης έκθεσης, μια που τόσος λίγος χρόνος κύλησε από την πρώτη έκθεση μέχρι σήμερα. Ε, και βέβαια υπάρχουν ένα σωρό σημεία στα οποία θα πρέπει να επανέλθουμε με την έκθεσή μας. Μια που έχουμε πρόσβαση σε πλέον στοιχεία, σε περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη, ε, επομένω θα πρέπει να το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα να ε, διαρθρώσουμε την έκθεση επίση. Θα πρέπει να δούμε με τους ηγητέ το πώ θα υπάρξει δυνατότητα να υποβληθούν κάποιες παρατηρήσεις και σχόλια πριν συντάξουν το κείμενό τους και έτσι να καλύψουμε και κάποια θέματα τα οποία τα συζητήσαμε στην πρώτη φάση, την αρχική. Και επίσης ελπίζω ότι στη διαδρομή αυτή της έκθεσης και με τις τροπολογίες θα αποφύγουμε το να μην έχει έκθεση ε, την προστιθέμενη αξία όσον αφορά το ύφος για κάποια τόσο σημαντικά ζητήματα. πρέπει να υπάρχει μετριοπάθεια βέβαια και από την μετριοπάθεια του ύφου προκύπτει η αξιοπιστία. Το είχαμε πει και για τους καταγγέλλοντες και είπαμε και για τη ΣΥΠΑ την περασμένη εβδομάδα οπότε και είδαμε ότι σε πολλά θέματα Υπάρχει δυσκολία στον αφορά την αποτελεσματικότητα, τη δικαιοσύνη σε σχέση με του καταγγέλλοντε, αλλά είναι βέβαια και θέμα δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Σιλβία. Έχουν δηλαδή και το θέμα των παρακρατουμένων φόρων και των επιστροφών. Αυτό μας είπε η Σιλβία είναι καλά μαντάτα. Επίση είναι πάρα το ότι αναφέρεται η ευκταία συνεργασία με τη ΣΥΠΑ που βρίσκει ανταπόκριση ιδίως από το Αμερικανικό Κογκρέσο και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, κάποιοι θεσμοί όπως το TTIP για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την καλή διακυβέρνηση. Επίσης να δούμε ποιος είναι, τι θα γίνει με αυτόν τον ελάχιστο αποτελεσματικό φόρο σε σχέση και με την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να συζητήσουμε τους συντελεστές και πάντως εγώ είμαι κατά αυτών των φόρων. Έχουν επισημανθεί τα προβλήματα σε σχέση με τον υπολογισμό αυτών των συντελεστών για τον ελάχιστο εφόρο τουλάχιστον αποτελεσματικό ανάλογα με τα κέρδη ανά χώρα φυσικά δεν μπορούμε το θέμα αυτό να το αφήσουμε απ' έξω από την έκθεση επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ελαστικοί στην έκθεση για το θέμα της απλούστασης του συστήματος και της αποτελεσματικότητάς του γιατί το ένα είναι απόρρια του άλλου. Επίσης, να αποφύγουμε τις τρευλώσεις και να πετύχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Διαφάνεια, να δούμε τι θα γίνει με το κόστος συμμόρφωσης. Οπότε όλα αυτά θα ξανασυζητηθούν και ενδελεχέστερα στην έκθεση από ό,τι έχουμε κουβεντιάσει μέχρι σήμερα. Τώρα, για τις ένομες τάξεις, τα κράτη τελικά που δεν συνεργάζονται. Θα πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος. Ό,τι μπορούμε πριν φτιαχτεί η μαύρη λίστα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και έτσι θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί σε αντίθεση με την κατάρτιση της μαύρης λίστας τώρα όσον αφορά με τις πληροφορίες για το beneficial ownership. Including, uh, there is a, point 45 uh, that calls for a global asset. Για τον τελικό κύριο ιδιοκτήτη είπαμε ότι εδώ πέρα μπορεί να υπάρξει ένα μητρό. Ναι, μακροπρόθεσμα με βρίσκει σύμφωνη κάτι τέτοιο. Αλλά βραχυπρόθεσμα η ανταλλαγή των πληροφοριών πριν φτιάξουμε αυτό το μητρό θα είναι χρήσιμη. Τέλο, νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιε ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Α πούμε το λέγει παράγραφος Δέλτα. Εκεί για τα δεδομένα. Και όλα αυτά είναι αφετηρία του να προχωρήσουμε και να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Ντανούντα, σε ευχαριστούμε, λέω πρόεδρε, ήταν πάρα πολύ ξεκαθαρό που είπε και τώρα ο λόγο στον ε, κύριο Λούγκε, ο οποίο αρνήθηκε να καθίσει εδώ στο Προεδρείο, παρά το ότι είναι αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι κάθισα στην αίθουσα γιατί θα μιλήσω ως και ο και όχι ως αντιπρόεδρος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, δύο εισηγητές. Ε, μπορώ να συμφωνήσω σχεδόν με όλα όσα είπε η Ντανούτα Χίμπνερ. Είναι νομίζω μια καλή ισορροπημένη έκθεση την οποία στο μεγαλύτερο μέρος την στηρίζω. Του του ε, θα ήθελα να αναφέρω τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η έκθεση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να φερθώ στη μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων. Εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς θα καταρτιστεί αυτή η λίστα, γιατί το ότι θα το κάνει η Κομισιόν σημαίνει ότι θα το κάνει κάποιος ο οποίος έχει διαφορετικά συμφέροντα. Π.χ. αν υποθέσουμε ότι ήταν η Τουρκία φορολογικός παράδεισος, δεν λέω ότι είναι, αλλά αν ήταν δεν θα την έβαζε στη μαύρη λίστα η Κομισιόν γιατί έχει και άλλα συμφέροντα. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε ε, πώς θα συνταχθεί αυτή η μαύρη λίστα και θα έπρεπε νομίζω να γίνει με, από κάποιον ανεξάρτητο ίσως από ένα επιστημονικό όργανο. Αυτό το οποίο δεν βλέπω εγώ στην έκθεση είναι ακριβώς μία αξιολόγηση του ρόλου των κρατών. Π.χ. λέμε εδώ πέρα πως δεν υπάρχει διαφάνεια από πλευράς επιχειρήσεων, αλλά τα εθνικά συστήματα φορολογίας, ειδικά εταιρική φορολογίας, ειδικά όσον αφορά την επιμέτρηση της ε, φορολογητέας ύλης, ε, δεν είναι και πολύ διάφανα. Π.χ. φαίνεται ότι δεν έχουμε σκεφτεί καθόλου το να απαγορεύσουμε τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις όταν ασκούν κάποια διακριτική ευχέρεια οι φορολογικές αρχές, είτε μιλάμε για transfer pricing, είτε για patent boxes, είτε για αποφάσεις που είναι στη διακριτική ευχέρεια των φορολογικών αρχών. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεση. Αυτό το οποίο επίσης ε, ε, είναι κάπως αρνητικό, είναι μια κάπως αφελής ερμηνεία για τον ρόλο των ε, τραπεζών. Παραδείγματο χάρη λέμε πώς θα μπορούσαν οι τράπεζες να είναι πιο συνεργάσιμες ε, για να μην μειωθεί η φορολογική βάση. Ε, δεν είναι αυτή η δουλειά των τραπεζών, αυτή είναι η δουλειά της εφορίας. Έτσι. Επίσης, δεν μπορεί να λέμε ότι οι τράπεζες ε, δεν θα πρέπει να στέλνουν χρήματα σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτή είναι η δουλειά των τραπεζών, να διασφαλίζουν τη ροή του χρήματος. Και πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Δεν είναι δυνατό να γράφουμε τέτοια πράγματα. Επίσης, όσον αφορά τον περιορισμό του ελευθέρου εμπορίου ως ένα μέτρο για να τιμωρηθούν τα κράτη-μέλη για τη φορολογική τους συμπεριφορά. Το ελεύθερο εμπόριο είναι κάτι από το οποίο αποφελούνται οι ιδιώτες και δεν είναι δυνατόν να ευθύνονται οι καταναλωτές και οι έμποροι για τη συμπεριφορά ενός κράτους. Οπότε δεν είναι δυνατόν, όπως είπα, όταν συμπεριφέρεται άσχημα ένα κράτος να τιμωρούνται οι παράγοντες της οικονομίας. Και επίσης, μετά την επίσκεψη στην ε, Ουάσιγκτον, τώρα αρχίζουμε να μπλέκουμε και την TTIP ε, στα φορολογικά πύχη. Κοιτάμε τα BEPS ε στο πλαίσιο του όσα υπάρχει σοβαρή αντίσταση, ειδικά από τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο για τα μέτρα BEPS. Αν το συνδυάσουμε αυτό με τα συναισθήματα των δημοκρατικών κατά του ελευθέρου εμπορίου, τότε ολόκληρη η TTIP πάει καλιά της, θα έλεγα. Λοιπόν, θα πρέπει να τα βλέπουμε ξεχωριστά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ε, έχω ακόμη τρία λεπτά, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ πέρα. Ευχαριστώ, Λούκε. Φίλιπ Λάμπερτς. Τι λέτε, εκτός μικροφώνου. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Φιλίππ είναι πάντα τόσο ευγενικό. τέλο πάντων, ξεκινάω με κάτι το θετικό. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, συνεισηγητέ που συνεργάστηκαν για όσα έγιναν που ήταν εξαιρετικά και τα τρία βασικά θέματα τα οποία θεώρησα τα θετικά της έκθεσης είναι τα εξή πρωτα Πρώτα-πρώτα, το θέμα για τους καταγγέλλοντες και την προστασία τους. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε επί τη βάση των όσων είχαμε στην πρώτη έκθεση συμφωνήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτών των πληρωμών και της ε, φορολόγησης στην πηγή. Αυτό είναι η ψήστη προτεραιότητα. Τότε που υπήρχε από την Ολλανδική Προεδρία εκείνη η ομάδα διοντολογίας, το είδε και η Επιτροπή, γιατί είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποια κενά στο φορολογικό δίκαιο. Επίσης, ήταν τολμηρή η σύσταση σε σχέση με την προτεραιότητά μας, δηλαδή να υπάρχουν κάποιο είδους αποτελεσματικές κυρώσεις που να θεσπιστούν. Ακόμα και να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, αν συνέτρεχε περίπτωση φόρο διαφυγής. Θυμάμαι στις συζητήσεις ε, της ΤΑΞ 1 ότι υπήρχε ε, η βούληση προς τούτο και είναι φυσικό εμάς που τώρα διαμορφώθηκε πλειοψηφία υπέρ. Πάντως παραθυράκια και κενά παραμένουν στο δίκαιο. Πρώτα-πρώτα. Διάβασα κάτι πολύ ενδιαφέρον σήμερα. Τα γαλλικά μου βέβαια δεν είναι και τα καλύτερα, αλλά έλεγε αυτή η εφημερίδα ότι η Βελγική ότι αρχίζουν κάποιο είδου επικοινωνίες προφορικές στο Λουξεμβούργο σε σχέση με φορολογικές ρυθμίσει. Εμείς φυσικά και πρέπει να τοποθετηθούμε Τώρα, όσον αφορά τη λίστα με τις φορολογικούς παραδείσους, πολύ σημαντικό. Όσοι έχουν πάει στη ΣΥΠΑ ξέρουν ότι όλες οι πολιτικές πτέρυγες θέλουν το ίδιο. Δηλαδή, ο, ο προηγούμενος επικεφαλής της Επιτροπής Φορολογών του, της Γερουσίας της ΣΥΠΑ έλεγε ότι από δημοτικής πλευράς αυτή η λίστα για τους παραδείσους φορολογικούς είναι ένας είναι μια, μια, μια κόλαση. Και λόγω αυτού του περίφημου beneficial ownership υπάρχει πρόβλημα και με τον Τέλαγο και, και είχαμε πει ότι στην έκθεση θα πρέπει να πούμε κάτι που να φυγραμμίζεται με αυτό το οποίο μας πρότεινε αυτός ο γερουσιαστής. Να μην έχουμε τη μαύρη λίστα, να μην έχουμε αναφορά χώρας προς χώρα. Γιατί βέβαια θα πρέπει να ονομάσουμε και παραδείσους και κάποιες αμερικανικές πολιτείες. Τώρα αυτά τα painted boxes. Εδώ να είμαστε πιο τολμήροι. Ήταν ξεκάθαρη τοποθέτηση του ΩΣΑ όπως διαπιστώσαμε στο Παρίσι αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών τον είπα ότι είναι εργαλεία για έρευνα και ανάπτυξη. Για το παρελθόν βέβαια δεν υπήρχε απόδειξη ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε. Εμείς πάντως θα πρέπει να δείξουμε τόλμη και να υποστηρίξουμε αυτή την ε, πρωτοβουλία. Ευχαριστώ τον Πίτερ που ετώνησε τα πιο σημαντικά. Αλλά με εξέπληξε το ότι η λιτότητα έχει τόσες συνέπειες που θα έπρεπε να πετάξει τον κάλαθο πολλά έγγραφα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε, δηλαδή και η δική μας Επιτροπή πόσο επηρεάζεται και τι θα κάνει. Μπάς και μπορεί η Επιτροπή να αποσπάσει κάποια πρακτικά από τις ενδιαφέρουσες συνεδριές του Συμβουλίου, γιατί έχουμε και κάποια άλλα έγγραφα. Εκεί που αναφέρεται ότι πρόκειται για μπερδεμένε καταστάσει, μπερδεμένα σκάνδαλα και επίση να δούμε τι θα γίνει με κάποια έγγραφα που έχουν παραπέσει, που έχουν σχέση και με το πλάνο Γιούγκερ. Οπότε, ας τα σκανάρει κάποιος, και εγώ μπορώ να το κάνω και να σας τα στείλω. Αυτό το λέω για την Επιτροπή. Ε, αν δεν ληφθούν όλα τα αναγκαία έγγραφα, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση. Ευχαριστούμε. Ανέφερες. Α, συγγνώμη, Λέω μιλητής, κάτι που ξεχάσαμε που δεν έχει να κάνει με την έκθεση. Το είπε βέβαια και ο Πίτερ ότι η περίοδος διαβούλευσης λύγει μέσα Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας τώρα που θέλουμε να πάρουμε τα έγγραφα. Πρόεδρος, αναφέρατε τις απροσδόκητες συνέπειες της λιτότητας, περιβαλλοντικές ανησυχίες της Κομισιόν έτσι θα δώσω το λόγο στο Φιλίπ Μα πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν. Ακριβώς αυτό ήθελα κι εγώ να πω. Να συνδέσω την οικονομία με τους φυσικούς πόρους. Αλλά μου τραβήξατε το χαλί κατά τα πόδια. θα συνεχίσω στα αγγλικά, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ τους δύο συνεισηγητές. Ελπίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε το δράμα που είχαμε σήμερα το πρωί. Θα δουλέψουμε επικοδομητικά μαζί σας για να πετύχουμε συνένεση, όπως και με το ταξένα. Τώρα, κάποια πράγματα που θα τονίσουμε στις τροπολογίες μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να τονίσουμε το τι μάθαμε από τα έγγραφα τα οποία πήραμε η παράταση της ταξέν είχε να κάνει με την πρόσβαση στα έγγραφα και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για το τι πήγε καλά, τι λειτουργήσε και τι όχι. κυρίω για το δεύτερο στην ομάδα κώδικα θεντολογίας. Τι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά την εντολή και τον τρόπο λειτουργία. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι κάποια στοιχεία μέτρησης επιβάλλονται κάθε φορά στις ίδιες χώρες δεν είμαστε τόσο ανόητοι να μην ε, αναγνωρίσουμε κάποιου είδους ε, καλούπι. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε την ανάλυση της παρακολούθησης των συστάσεων Tax 1. Θυμάμαι εξάλλου ότι ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι για την προστασία των καταγγελόντων μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Φτάνουμε στον Ιούνιο του 2016 και εγώ δεν βλέπω τίποτα και ειλικρινά όταν άκουσα την αντίδραση της Μαριάν Τάισεν εκ μέρου της Επιτροπής στην Ολομέλεια της Προάλλες, πραγματικά με εξέπληξε, ήταν στο το παράδεκτο, είναι κάτι που δεν μπορώ να στηρίξω. Ανάλυση του ρόλου των ευρωπαϊκών χωρών επί των εξαρτημένων τους ε, επικρατιών, εδαφών. Κάποιοι παίζουν παιχνίδια με μας. Λένε, ναι βεβαίως, αλλά στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη φορολογική παράδειση που έχουμε στην Ευρώπη. Πρέπει να τονίσουμε υπόψη και το θέμα των ερευνών που γίνονται για τις κρατικές επιδοτήσεις, γιατί είναι εξοργιστικό από τις τρεις χώρες μέλη που καταδικάστηκαν μόνο μία άνοιξε ένα λογαριασμό για να πληρωθούν τα χρήματα. Το Βέλγιο και κάτω χώρες εξακολουθούν να μην εισπράττουν τα χρήματα. Κάτι που είναι απαράδεκτο, γιατί δεν είναι επειδή πήγε στο δικαστήριο που δεν πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση της Επιτροπής καθόλου. Πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση και πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό και να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο Φάμπιο για το ρόλο των ενδιάμεσων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζών, ε, δικηγορικών γραφείων κλπ. Πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό που πιστεύουμε, δηλαδή να προτείνονται κυρώσεις. Τώρα για τα διάφορα boxes για την έρευνα και την ανάπτυξη κλπ. Αν θέλετε να ενθαρρύνετε την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, αυτό το κάνετε με απευθείας ε, επιδότηση, αλλά όχι με εξαιρέσεις φορολογικού τύπου. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά τα patent boxes πρέπει να καταργηθούν το αργότερο μέχρι το 2020. Και έπειτα Κάτι που συχνά βλέπουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Διαπιστώνουμε, σημειώνουμε, παρατηρούμε, θα που. Εγώ νομίζω ότι πρέπει η διατύπωσή μας να είναι πιο έντονη. Είναι σοβαρές υποθέσεις αυτές. Βλέπουμε την απογοήτευση των πολιτών. Αν θέλουμε να δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε το θυμό τους, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε, αν όχι θυμωμένο λόγο, τουλάχιστον πιο έντονο λόγο, ότι απαιτούμε να αλλάξουν τα πράγματα και όχι ότι ε, εκτιμούμε, λάβετε υπόψη σας αυτά που κάνουμε. Όχι, να είναι πιο οξύ ο τόνος μας. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που είχα να κάνω. Νομίζω πέντε λεφτά κράτησε η παρουσίασή μου. Πρόεδρος, συγχαρητήρια και για το περιεχόμενο και για την πειθαρχία που επιδείξατε. Πράγματι, εσείς συζητάτε πιο πολιτικό τόνο και λιγότερο διπλωματικό. Ωραία, θα το συζητήσουμε, αλλά μια παρατήρηση τώρα που μου έρχεται στο μυαλό ακούγοντάς σας. Ότι σε ένα χρόνο με τη τάξη 1 και τη τάξη 2 καταφέραμε να επιδείξουμε την αξιοπιστία μας, την πολιτική αξιοπιστία μας. Επίσης, τις ακροάσεις που κάνουμε, είδαμε εντάξει, όσοι δεν θέλησαν να έρθουν, οι πολυεθνικές τράπεζες κτλ, τις ξέρουμε και στις διακυβερνητικές διασκέψεις που οργανώσαμε, ακούσαμε επίσης πολλούς. Είχαμε τέσσερις διακοινοβουλευτικές μέσα σε ένα χρόνο με τα κοινοβούλια των 28 χωρών μελών και θα θυμόσαστε ότι στην πρώτη συνάντηση πολλοί είπαν ήρθαμε αλλά αναρωτιόμαστε γιατί ανακατεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή την υπόθεση. Και μετά την τρίτη συνάντηση οι ίδιοι μας λέγανε είναι πολύ σημαντικό πρέπει να συνεργαστούμε και ευχαριστούμε για την οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Και όσοι ήρθαν στις Ηνωμένε Πολιτείε διαπίστωσαν ότι ούτε στο Κογκρέσο, ούτε στη Γερουσία, ούτε στη Βουλή των Αντιπροσωπών, ούτε οι Δημοκράτε, ούτε οι συντηρητικοί, κανένα δεν αφισβήτησε την ε, πολιτική δυνατότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί από αυτών των ζητημάτων. Θεώρησαν ότι είναι απολύτω ε, θεμητό, κανεί δεν το αφισβήτησε είπανε ότι είναι ευτυχείς που έχουν έναν Ευρωπαίο συνομιλητή που μιλάει εκ μέρους της Ευρώπης και μάλιστα τονίζοντας και που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας, είτε μεταξύ των χωρών μας, είτε μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών εδώ. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας. Και όπως λέει και ο Φιλίπ Λάμπερτς, ακριβώς αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να προφέρουμε πολιτικό λόγο. Τώρα, το λόγο έχει ο Ντέβιτ Κόμπερν για το EFDD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό και να μην το κάνετε για τη Μεγάλη Βρετανία. Θα έχουμε φύγει εμείς. Αλλά η έκθεση αυτή ζητά από την Κομισιόν ε, να φέρει μια κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων. Πολύ κακή ιδέα θα γίνουν οι επιχειρήσεις λιγότερο ανταγωνιστικές και θα αυξηθεί το μέγεθος του κράτους. Η εναρμόνιση των εταιρικών φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί βεβαίως ε, να είναι λογική για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά ο πραγματικός στόχος είναι να αυξηθούν οι φόροι. Μην ξεχνάμε πως τελικά οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερο. Το κόστος θα το περάσουν στους πελάτες οι επιχειρήσεις οι χώρες όπως η Σοσιαλιστική Γαλλία με υψηλούς φόρους δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με χώρες ε, όπως τη Μεγάλη Βρετανία που έχουν χαμηλούς εταιρικούς φόρους ή την Ιρλανδία. Η λύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταστρέψει αυτός που είναι παγκοσμίω ανταγωνιστικοί. Και αν χώρες σαν την Βρετανία θέλουν να έχουν ένα παγκοσμίω ανταγωνιστικό περιβάλλον για να δημιουργούν δουλειές και πλούτο όπως κάνουμε τότε πρέπει να φύγουμε από την Ένωση που στόχο έχει να ελέγξει τη φορολογία. Επίσης η έκθεση καροσολίζει το πακέτο αποφυγής της φορολογίας. Τα συστήματα τα φορολογικά της Αγγλίας και της Σκοτίας επερίπτουν ευθύνη στους ε, διευθυντές των εταιριών να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν απέναντι στους μετόχους για να μειωθεί ο φόρος. Οι γενικοί κανόνες κατά της φοροαποφυγής, όπως ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ερμηνευτούν δύσκολα και ο στόχος είναι να τρομοκρατηθούν οι απλοί φορολογούμενοι. Δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά των μεγάλων επιχειρήσεων όπως λέτε, αλλά κατά των ατόμων εκείνων που δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρους για να τα αποφύγουν. Το καλύτερο είναι ένα απλό φορολογικό σύστημα, έτσι ώστε ο απλός φορολογούμενος να ξέρει πόσο έχει να πληρώσει. Αντί να καταλήξουμε σε αυτούς τους κανόνες για να πληρώνει ο απλός φορολογούμενος περισσότερους φορούς σήμερα, καταψήφισα και προσπάθησα να σταματήσω την Επιτροπή από το να βγάλει ευρωπαϊκό αφημί. Ξέρουμε προς τα που πηγαίνετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως δεν θα το πει πριν από το δημοψήφισμα, αλλά θέλετε να φορολογήσετε τους Βρετανούς απευθείας, εάν παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, προτείνεται εδώ πέρα πανευρωπαϊκό φόρο στην πηγή και ένα κέντρο συντονισμού. Ευρωπαϊκή δόη δηλαδή. Και τι άλλο ένα γενικό αρχείο όλων των στοιχείων ενεργητικού των εταιριών. Οπωσδήποτε όλα αυτά εν ώψη ενός πανευρωπαϊκού φόρου πλούτου. Όλα αυτά θα ενισχύσουν τον Brexit και εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να ενημερώσω τους Βρετανούς πολίτες, τους εργατικούς που θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους ε, έτσι ώστε να τα ξέρουν. Πρόκειται για πράγματα αποκρουστικά και αυταρχικά και ελπίζω πραγματικά να σηκωθούμε, να φύγουμε και να γλιτώσουμε από αυτές τις αηδίες. If αυτή την περίπτωση θα μας λείψετε. Θα σας λείψουν τα λεφτά μας. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Με το ευρώ εκεί πέρα που έχετε κολλήσει. Speak to a French about EU money. μιλάτε σε έναν Γάλλο για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ένα δισεκατομμύριο ευρώ πληρώνουν οι Γάλλοι για τη συνεισφορά. Εκτός μικροφώνου. Μπερνάρ Μονό από το ENF. Δεν θα μιλήσω για Frexit. Κύριε Σιγητά, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την ποιότητα του έργου σας. Γνωρίζετε ε, πόσο η ομάδα μας είναι υπέρ της κυριαρχίας ε, των ε, χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αντικαταστήσει τις κρατικές αρχές. Εδώ μιλάμε για πραγματική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον υπάρχει μια ενιαία αγορά με ελευθερία κυκλοφορία κεφάλων. Το LuxLeaks, το Panama Papers, οι πρακτικές, οι φορολογικές της Apple, της IKEA, Starbucks κλπ. μας αναγκάζουν να αντιδράσουμε με δύναμη η ομάδα μας ήταν υπέρ της έκθεσης TAX 1 και πάντα συμφωνούσε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της απάτης και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Με τις τέσσερις εκθέσεις που ε, καταρρύπτουν το απόρριτο Ελβετίας, Λιχνεστάν και τα λοιπά. Συμφωνήσαμε και σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την εφαρμογή 6 μέτρων κατά της ε, φόρο αποφυγής μέσω της ΑΠΑΤ. Όμως με την έκθεση τάξη 2 προβληματίζομαι. Δεν είχαμε κάποια έγγραφα, έπρεπε να περιμένουμε περισσότερο, ε, δεν ήρθαν διάφοροι να μας μιλήσουν για σκάνδαλα, τετράπεζες, τα άλλες δικαιοδοσίες. Τα Panama Papers έδειξαν ότι πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας. Οι απόλυτα θεμητές προσπάθειές μας δεν πρέπει με τίποτα να αποτελήσουν το άλοθη για μια φορολογική ένωση. Είμαστε κατά. Συνεπώ, θέλω αυτή την κόκκινη γραμμή να την θέσω και πάλι όσον αφορά την ομάδα μα. Ενώ το σημείο 38 της σα, σε ένα μεγάλο βαθμό, ακριβώ είναι όσων πιστεύουμε εμεί, οι πατριώτε. Με τίποτα δεν θέλουμε, εκτό βέβαια αμφισβητηθεί η ομοφωνία, ένα ανεξάρτητο όργανο της Επιτροπής να έχει πολιτικό έλεγχο στα φορολογικά των χωρών μελών. Έτσι το παρουσιάζετε εσείς. Πάντως χαιρετήσω την προσπάθεια του εισηγητή που την ευθύνη τη ρίχνει στο Συμβούλιο. Γιατί είναι αλήθεια ότι την ευθύνη των, η ευθύνη των ενδιάμεσων στα σκάνδαλα που γνωρίζουμε είναι τεράστια. Κάνουν lobbying στην Επιτροπή και το Συμβούλιο για να βγουν λάδι. Εμείς όμως πρέπει να αντισταθούμε. Θα προτιμούσα κυρώσει σε όσους έχουν βοηθήσει την φοροαποφυγή, είτε πρόκειται για δικηγορικά γραφεία, είτε σε βούλους είτε άλλους. Και θέλω προστασία των καταγγελόντων. Ακόμα και αν η Γαλλία έχει ήδη νομοθετήσει γι' αυτό, θα ήθελα και η Ευρώπη να το κάνει. Η ανησυχία μου είναι ότι αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή σε νέε πρακτικέ, οι οποίε προσπαθούν να παρακάψουν του κανόνε που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ τι πρακτικέ πρέπει να τι καταργήσουμε και να είμαστε σε γρήγορε να προσέξουμε πάρα πολύ όσον αφορά τώρα τη φορολογική ηθική μεταξύ των φορολογουμένων για τα διαφυγόντα κέρδη. Πρέπει να ανακτηθούν τα ποσά αυτά και οι εθνικές φορολογικές αρχές πρέπει να είναι αδιάλακτες. Η τελική έκθεση θα πρέπει να το συστήνει αυτό. Καταλαβαίνω ότι Google εποφελήθηκε, όμως είναι σαν να πρηματοδοτούμε την απάτη. Τέλος. Προσθέτω ότι όλα, όλος ο προβληματισμός μας πρέπει να μπει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που να δείχνει την τρελή κατάσταση όσον αφορά τις κρατικές δαπάνες. Γιατί, Γιατί οι χώρες χρηματοδοτούν τις πολιτικές τους που είναι υπέρ του προπολογισμού βασικά και τίποτα άλλο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο να χειριστούμε τον προπολογισμό μας να τιμωρηθεί κάθε, κάθε τρόπος φοροποφυγής και φοροδιαφυγής και γι' αυτό πρέπει να επανέλθουμε σε ποσοστά εισφοράς που να είναι συμβατά με την επιχειρητικότητα. Περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσβλέπω στη συνέχιση των διαβουλεύσεών μας. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μια που όλοι τηρείται το χρονικό όριο, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο θα δώσουμε σε τέσσερις το λόγο, τρία λεπτά καθώς και ξεκινούμε από τον Γκούναρ Χέκμαρ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα. Συμφωνώ πρώτα με την απόψή σας ότι μία από τις πιο εντυπωσιακές συνέπειες του Brexit είναι ότι θα μας λείψουν κάποιες προσωπικότητες όπως ο συνάδελφος που έλαβε πριν το λόγο. και αισθάνομαι πολύ θαραλέος όταν περιγράφω το πόσο φρικτά είναι τα πράγματα εδώ που βρισκόμαστε, έτσι είναι. Σας αρέσει η περιπέτεια σε εσάς τους Βρετανούς, αλλά εδώ είμαστε τέλος πάντων. Οπότε, να, θα μας λείψετε άμα γίνει το Brexit. Εγώ ελπίζω να, να μείνετε και να ακούμε κάποιους σας και να μας ε, ε, κάνετε να ακουγόμαστε ως πολύ μετριοπαθή. Πάντως ευχαριστώ τους συγητές και θέλω επίσης να αναφέρω ότι όταν μιλούμε για φορολογικά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μας διακρίνει ακρίβεια. Πρώτα πρώτα. Δεν είναι δυνατόν να ζητούμε νομοθεσία που να τιμωρεί αυτούς που τηρούν τον νόμο γιατί κάποιες σχετικές προτάσεις προσπαθούν να κηρύξουν παρανόμους τους νομιμόφρονες. Δεν γίνεται έτσι στο κράτος δικαίου. Θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η απάτη για τα φορολογικά, η ποινικά κολλαζόμενη ε, φοροδιαφυγή και άρα θα πρέπει η νομοθεσία μας να είναι τέτοια ούτως ώστε να κλείνει τα παραθυράκια και τα αέρητα κενά του νόμου. Αλλά όλα να ανακοινούνται στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Επίσης, με εξέλιψαν κάποια σημεία συζήτηση αλλά και του κειμένου γιατί αναφέρεται κάπου, υπάρχει το πνεύμα ότι είναι ζαβολιάριδε οι επιχειρηματίε στην Ευρώπη και δεν πληρώνουν του φόρου του. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ούτε είναι σωστό τρόπο ούτω ώστε κάποιο να μπορεί να ελκύσει ε, επενδύσει και να δημιουργήσει θέσει εργασία στην Ευρώπη. Ούτε ισχύει ότι αλλού είναι χαμηλότερη φορά. Να μην ξεχνούμε ότι εμείς έχουμε 10-15% ε, περισσότερους φόρους από ότι ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι οι πολυεθνικές βεβαίως και θα τους αρέσουν αυτές οι λύσεις. Εντάξει, έτσι είναι η αγορά. Ανταγωνισμός. Όμως, ας εξασφαλίσουμε το ότι εμείς θα τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τι φορολογικές ρυθμίσεις για να διαπράξουν το έγκλημα της φοροδιαφυγής. Μην ξεχνούμε όμως εδώ πέρα οι φόροι είναι οι πιο υψηλοί στον κόσμο εδώ στην Ευρώπη. Επομένως, να δούμε πώς δεν θα υπονομεύσουμε τις εθνικές αρμοδιότητες και ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προσέξουν την εφαρμογή των όσων θα θεσπίσουμε για να μην δημιουργηθούν καινούργια παρατηράκια και κενά στο δίκαιο. και προσοχή να μην δυναμητήσουμε επίσης την παγκόσμια ανάπτυξη με τα όσα λέμε για ελεύθερο εμπόριο. Πέτρα Τζίμον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τους συζητητές ε, το σχέδιο έκθεσης ε, που ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα που έχουν μείνει από την τάξη. Ε, νομίζω πως είναι σημαντικό να πούμε πως το σχέδιο έκθεσης για τους ε, καταγγέλλοντες είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθει σοβαρά υπόψη. Επίσης αναφέρθηκε το τι θα γίνει με την ευνοϊκή μεταρρύθμιση των ευρεσιτεχνιών, τα λεγόμενα patent boxes. Κοιτάξτε, είχαμε μια συνεδρίαση στο Παρίσι με τον ΟΣΑ και η σαφήνεια με την οποία ο ΟΣΑ λέει πως κατά την άποψή του θα πρέπει επί της αρχής να καταργηθούν ε, τα patent boxes και να προωθηθεί η έρευνα και ανάπτυξη με τρόπο που δεν θα βλάπτει τη φορολογία και εμείς δεν ξέρουμε ακόμη το τι θα κάνουμε με αυτά ενώ πρέπει να καταργηθούν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να συνοηθούμε να κάνουμε μια κοινή μαύρη λίστα που θα περιλαμβάνει και κράτη-μέλη. Και οπωσδήποτε θα έχουμε συναρπαστικές συζητήσεις. Επίσης εγώ το εξής θα πω. Ναι, ρητορικά γίνεται αυτοί δηλαδή οι οποίοι βλάπτουν περισσότερο τον φορολογούμενο να λένε ότι προστατεύουν τους στοχούς. Ότι γίνεται ρητορικά από τη μία να λέμε ότι αποφεύγουμε φόρους ε, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Είναι λανθασμένο ε, είναι οπωσδήποτε φρασίτατο, αλλά τουλάχιστον είναι ρητορικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Πήρε τον λόγο εκ νέου στον Μπέντ Λούκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Το ένα αφορά τη φορολόγηση στην πηγή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ε, γιατί εδώ πέρα εννοείται έναν ευρωπαϊκό φόρο. Δεν υπάρχει νομική βάση. Ε, νομική βάση υπάρχει μόνο για 28 εθνικούς φόρους στην πηγή. Βεβαίως αυτό δεν προωθεί τη διαφάνεια. Θα πρέπει απλά να κλείσουν τα παραθυράκια στην εθνική φορολογική νομοθεσία που δίνουν την δυνατότητα να ε, σκεφτόμαστε τη φορολόγηση στην πηγή. Επίσης, απαιτούμε εδώ πέρα μια ελάχιστη ε, πραγματική φορολογία. Και πάλι αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαίωμα να μπει σε αυτό το ζήτημα. Είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Οπότε και εδώ πέρα είμαστε επικριτικοί, όπως και στην απαγόρευση των patent boxes. Όλα αυτά είναι εθνικές αρμοδιότητες. Οπότε η ευνοϊκή μεταχείριση των ευρεσιτεχνιών είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετο Το είπαν και άλλοι, είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την πρόθεση της έρευνας και της ανάπτυξης. Επίσης, προτείνεται να υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Συνοχής ε, και Συντονισμού. Και πρόκειται εδώ πέρα για μια νέα αρμοδιότητα η οποία δεν ε, υπάρχει. Θα πρέπει το πολύ πολύ να ενισχυθούν ε, οι αρμοδιότητες της ομάδας επαφής για να γίνουν αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ. Και τέλος, δύο πράγματα στα οποία φοβάμαι πως ε, έχει μπει εδώ πέρα πραγματικά ο Ταύρος στο Ιαλοπολείο. ένα μητρό όλων των περιουσιακών στοιχείων που έχουν άτομα και εταιρίες και καταπιστεύματα και ιδρύματα στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές. Αυτό θα ήταν ένα καλό μέτρο για να τρομάξουμε το κεφάλαιο και να μην ξαναέρθει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πως το κεφάλαιο είναι πολύ ευέλικτο και ευκίνητο. Και έχει και άλλες δυνατότητες για να ε, χρησιμοποιηθεί παραγωγικά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. στις ΗΠΑ έχει ξεκαθαρίσει το ότι το θεωρούν προσβολή το να λάβουμε μέτρα κατά της ΜΠΕΠΣ στο πλαίσιο του ΩΣΑ και θα μπορούσε να επηρεαστεί και η θέλησή τους να συζητήσουν τέτοια μέτρα. Βέβαια, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί με τον ζήλο που έχουμε για αυτά τα μέτρα κατά της BEPS. Ε, Όχι γιατί επειδή είναι επί της αρχής ε, λάθος, αλλά γιατί κλείνουμε πόρτες που θα έπρεπε να έχουμε ανοιχτές, εάν θέμε να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή. Ευχαριστώ και για τον χρόνο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Εμείς ε, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρος που θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο για να απαντήσουν οι συντάκτε ή ο συντάκτη. Τελευταίο ήταν και σορτάσουν ε, για του Πρασίνου. Συγγνώμη οι άλλοι, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ορτάσουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα πω κάτι ε, επιπλέον των Ισπανική Λαμπετσάρη. Έχουμε και το σημείο 30, το οποίο 30 για του καταγγέλτε είναι πάρα πολύ βασικό. Ευχαριστώ είναι πολύ σωστό, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνούμε, του εισηγητέ τέλο πάντων, ότι αυτό το οποίο σου κάνει την γνώμη είναι ότι όσα έχουν κάνει με του φόρου είναι πολύ σημαντικά. Επομένω, θα πρέπει το κοινοβούλιο να είναι κατηγορηματικό σε όσα θα πει αντίστοιχα. Κάτι άλλο για τι αποστολέ και σε Κύπρο και σε είπα. Είδαμε ότι υπάρχουν θέματα ξεπλήματος χρήματος. Άρα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το φαινόμενο. Δεύτερον, όσον αφορά την blacklist τρίτων χωρών, ε, ήδη αναφέρθηκε, αλλά εγώ σας το τονίζω ότι αυτή η λίστα δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε ανταλλαγή των πληροφοριών, αλλά θα πρέπει επίσης να αφορά και τους φορολογικούς παραδείσους. Τρίτον, σχέση φορολογίας και συμφωνίων ελευθέρου εμπορίου. Υπάρχει μια ρήτρα στην που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα χρηστή διακυβέρνηση σε κάποια συμφωνία εμπορική. Ε, θα πρέπει να κάνουμε όμω το παραπάνω βήμα. Να έχουμε δηλαδή κάποιο κατάλογο ε, σημαντικών ε, προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρούνται και έτσι να εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει αυτόματη ε, ανταλλαγή πληροφοριών με την χώρα με την οποία θέλουμε να κλείσουμε μια συμφωνία. Τέλος, Όσον αφορά τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ολομέλειά μα επανειλημμένα έχει ζητήσει από την ΕΤΕ να μην συνεργάζεται με τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα, ειδικέ φορολογικέ ένομε τάξει και κράτη. Η πολιτική μας ομάδα, κύριε Πρόεδρε, θα υποβάλει τροπολογίες σε σχέση με αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ. Εμεί εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Άντε, θέλετε. Όχι κάτι ενημερωτικά, θεωρώ. Ότι είναι αντισυνταγματικό το να γίνεται έλεγχος της περιουσίας των ιδιωτών. Αυτό ισχύει στην ε, Βρετανία. Μπορεί στην Ευρώπη να το κάνετε, στη χώρα μας όμως όχι. Σίγουρα και θα υπάρξει βέτο αν θέλετε να περάσετε κάτι τέτοιο, αν είμαστε στην Ευρώπη. Το πρόβλημα με τη Βρετανία, λέει ο Πρόεδρος, είναι ότι δεν υπάρχει όμως γραπτό σύνταγμα. Όμως όταν εσείς είχατε δικτατορία, εμείς δεν είχαμε. δεν ήθελα να επικρίνω την Βρετανική Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος. Ελπίζω, ελπίζω, λέει ο ο αγορητής. Κύριε Ισηγητά, τι συμπέρασμα βγάζετε από όλη αυτή την πλούσια κουβέντα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα πρώτα για την κυρία Χούμπνερ. Την ευχαριστώ και εγώ να τονίσω αυτά τα οποία είπε για τους ε, καταγγέλλοντες. Θα πρέπει να τα πούμε κατηγορηματικά και <clears throat> στα ράτα. Άρα θα ασχοληθούμε με αυτό. Όσον αφορά τη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, Πήγαμε κάποιοι από εμά την περασμένη εβδομάδα στη ΣΥΠΑ και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την ε, Φορολογική Επιτροπή. Άρα θα πρέπει ε, όλα αυτά να τα καλύψουμε. Να είναι δηλαδή παγκόσμια η αντιμετώπιση. Έτσι θα είναι πιο θεμητιόρη του παιχνιδιού. Πιο δίκαιη. Τα είπαμε το Κογκρέσο, τα είπαμε με την κυβέρνηση. Ε, είμαστε στην αρχή μόνο τη συνεργασία μα για τον κύριο Μπέρντ Λούκε. Δεν υπάρχει να καλύψω όλα όσα είπε, αλλά πάντως έχουμε πάει περισσότερο επενδυμένα στον ΩΣΑ. Και τα patent boxes και τα συναφή δεν συνάδουν με μια καλή οικονομική πολιτική, είπαμε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο για τις επενδύσεις. Αν κανείς θέλει να έχει τα ίδια αποτελέσματα, αντί για φορολογικά κίνητρα και ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις, ας δίνει ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Συμφωνώ δηλαδή μαζί σας, κύριε Λούκη. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση για το Μητρό, όσον αφορά τα περισσότερα στοιχεία. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί θέλουμε να είναι προβληματικό αν η φορολογική αρχή έχει πρόσβαση σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν κάποιο είναι νομιμόφρον ω νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Πληρώνει το φόρο που του αναλογεί. Αυτό θα ενοχλούσε μόνο αυτούς που έχουν κάτι να κρύψουν από τις φορολογικές αρχές. Απαράδεκτο. Άρα μάλλον διαφωνώ μαζί σας. Τώρα όσον αφορά τη Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου, τα έχουμε συζητήσει αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε ότι κάποιες ε, εταιρείε έχουν εκμεταλλευτεί αυτές τις συμφωνίες για να παρανομήσουν. Προσωπικά θέλω να υπάρχει περισσότερο δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον οι μεγάλες εταιρείε να πληρώνουν τους φόρους τους. Άρα, υπάρχει εξωτερική διάσταση στο θέμα της καλής διακυβέρνησης, στο θέμα της βολογικής πολιτικής. Οπότε ίσως σε αυτό το σημείο διαφοροποιούμαστε. να συνεργαστούμε. Τώρα για τους καταγγέλλοντες, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό σημείο. Να το δούμε. Φάμπιο, ευχαριστώ για τόσα είπες. Θα τα συζητήσουμε, σίγουρα. Και για τον Φιλιπ Λαμπέρ έχω να πω, α, έχει φύγει ο Φιλίπ, αλλά πάντως και αυτός ανέφερε για τους καταγγέλλοντες. Και εκεί θα πρέπει να τα πούμε σταράτα και για τα patent boxes. Συμφωνούμε. Τώρα σχετικά με Βέλγιο και κάτω χώρες. Συνεχίζουν ε, κάποια αρνητικά σημεία παρά τις αποφάσεις της Επιτροπής για τις φορολογικές ρυθμίσεις. Και τα είπαμε και στην πρώτη έκθεση ότι η ανάκαμψη μετά την απόφαση της Επιτροπής το να καταβληθεί κάποιος φόρος αποτελεί κάποιο παράδοξο. Γιατί έτσι ενθυλακώνει τα χρήματα η χώρα που είχε θεσπίσει τα στραβά. Θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Πριν μας είπατε για το φορολογικό πακέτο, αλλά σήμερα ε, είχατε απόσχη. Άλλα μας είπατε τώρα και άλλα κάνατε το πρωί. Έτσι βλέπω. Δεν ξέρω, τόσο αν δεν κατάλαβα καλά τα όσα μας είπατε. Θα έπρεπε τα σχετικά μέτρα να τα υπερψηφίσετε το πρωί, δεν το κάνετε. Τέλος πάντων πολλά και ενδιαφέροντα αναφέρθηκαν και σε συνεργασία με τον κύριο Τόιρερ θα καλύψουμε τα όσα είπατε στην έκθεση, θα τη βελτιώσουμε και θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά και τελικά να έχουμε μια αξιόλογη έκθεση. Δεν έχω τα 5 λεπτά, όντως. Αλλά σας αναφέρω πώς. Θα πρέπει να γίνει ευρύτερη συζήτηση όσον αφορά τη φορολογική πολιτική και αυτό είναι θέμα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά υπάρχει η ενιαία αγορά. Έχουμε ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Πρόκειται για συνεργασία μα. Άρα θα πρέπει όσον αφορά τη διαφάνεια, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη φορολογία και τη συνεργασία χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνε. Αυτά όλα είναι και Είναι αλληλεξαρτώμενα οπότε Γι' αυτό και εργαζόμεθα εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ακριβώς όπως έγινε και με την τάξη ένα έφυγε η κυρία Φερέρα ε, η οποία ήταν στην αρχή εδώ, αλλά ε, για την πρώτη έκθεση δούλεψε η κυρία Φερέρα και ο κύριος Τόρερ που δεν είναι εδώ. Θα πρέπει να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ τόλμης και αποτελεσματικότητας. Έχει ε, ο κύριος Λαμπέρ σε σχέση με το πόσο διπλωματικοί θα πρέπει να είμαστε. Να είμαστε ρεαλιστές επομένω. Μόνο έτσι θα πιάσουν τόπο αυτά τα οποία λέμε. Έτσι θα ελκύσουν μόνο την προσοχή για όσα λέμε και θα ε, μας ακούσει ο κόσμος. Πλατείας πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΩΣΑ, ε, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κογκρέσο, είχαμε επαφές με όλους αυτούς και είναι διπλή η δική μου εντύπωση ότι υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει και πολιτική υποχρέωση ούτως ώστε το θέμα να προχωρήσει υποχρεωτικά και να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την καταπολέμηση των παρανόμων ε, πρακτικών και των ε, καταχρηστικών νομοθεσιών. Αυτό είναι υποχρέωση του πολιτικού κόσμου. Ταυτοχρόνως δε έχω την εντύπωση ότι η πρόταση ΟΣΑ είναι μέση οδός. Δεν συμφωνούν όλοι. Άλλοι θέλουν ότι είναι τόσο τολμηροί, άλλοι θέλουν ότι είναι υπερβολική. Η τελικά, παγκοσμίω θα καταφέρουν τα κράτη να συμφωνήσουν σε κάτι που θα προσωμιάζει με την πρόταση του ΩΣΑ. Οπότε έχουμε μια πρόταση και εμείς επίσης θα κάνουμε άλλη πρόταση, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η δεύτερη έκθεση, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει αυτό το στοιχείο, το αξιολογικό, παρά το ότι δεν συμφωνούν όλοι. Και επίση ε, έχει σημασία και το εξή Από τότε που ξέσπασε η υπόθεση των Panama Papers έχει δοθεί μια όθηση εκ νέου στο θέμα και εκφράζεται σε επίπεδο κρατών, σε επίπεδο κυβερνήσεων. Έχουμε την Σάντζη Κορυφή του Λονδίνου. Και στο περιθώριο αυτό, σημαντικές χώρες είπαν ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό του πραγματικού δικαιούχου, του beneficial owner. Οπότε οι χώρες, οι όμιλοι εταιριών θα πρέπει να παρέχουν υποχρεωτικά κάποιες ε, ε, πληροφορίες ή να δημοσιοποιούν το ποιος είναι ε, ο πραγματικός δικαιούχος Οπότε έτσι δόθηκε στην υπόθεσή μας μια όθηση. Αυτά λέω που μας απειλούν στο ταξένα και που μας απασχολούν τώρα. Οπότε είπαμε ότι αυτό το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε είναι ε, ορόσημο, είναι σημείο κλειδί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια εύστοχη δόκιμη λύση, χωρίς να είμαστε ε, κατά της ε, επιχειρηματικότητας ή της ε, ανάπτυξης, αλλά θα βοηθήσουμε να υπάρχει υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού, να την δικαιοσύνη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Τώρα κάτι άλλο επίσης ότι αυτή την ώρα, αυτή την ώρα στο Παρίσι έχουμε δεκάδες ε, υπαλλήλους του γαλλικού ΣΔΟΕ τέλος πάντων και οι οποίοι εισέβαλαν ε, για να κάνουν ευθυντικούς ελέγχους στο γαλλικό Google για να δούνε κατά πόσον ε, συμμορφώνεται το γαλλικό Google με το γαλλικό φορολογικό δίκαιο. Μας έχουμε όλες αυτές τις ε, πρωτοβουλίες και οπότε και εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε την πιο δόκιμη, την πιο σωροπή λύση αυτή είναι η δουλειά μας. Οπότε για να δούμε τώρα το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας. Έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά τις συνεδριάσεις ε, που αφορούν τη συνάντηση των σκιωδών και των ε, ε, βασικών των εισηγητών. Τα έχετε αυτά λάβει στο φάκελο. Μιλάμε για τις 2 έκτου έξω στο Στρασβούργο, 7, 9, 13 και ενδεχομένως και στις 15. Η δεκαταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες Είπαμε μετατίθεται για τι 31 Μαου επομένω έχουμε μια εβδομάδα παραπάνω, το μεσημέρι θα έχω στις πρώτες και οπότε εγώ το έχω σημειώσει ότι θα γίνει ό,τι μπορούμε, θα το πούνε και οι συντονιστέ, ότι θα, ε, έτσι θα έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε τα έγγραφα που διάθεσή μας, αλλά και όσα θα, θα, θα, θα μπορέσουμε να ε, έχουμε στα χέρια μα. οπότε θα γίνει η συζήτηση στην Επιτροπή μας στις 21 ε, Ιουνίου, όπως συμφώνησαν οι συνεισηγητές και κατόπιν θα ακολουθήσει ε, η εξέταση από την Ολομέλεια. Είμαστε ήδη στις 4.30, δύο λεπτά και διάλειμμα, ώστε να ε, έρθει η πρόεδρος Μακαβάν αλλά και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ανάπτυξης για την υπόλοιπη